Pasemos al debate sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el reglamento. Έχουμε τη σύσταση του τροποποιητικού κανονισμού 1234-2007 όσον αφορά την κοινή οργάνωση αγορά, όπου έχουμε κάποιε συγκεκριμένε διατάξει για συγκεκριμένα προϊόντα. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει το λόγο η Επίτροπο, η κυρία Φίσλερ. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που δώσατε το πράσινο φως στην επίγουσα διαδικασία. Ελπίζω έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο ε, την κατάσταση. Τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο γαλακτοκομικός τομέας. Μία λύση να ενταχθεί το γάλα στο άρθρο 186 και η άλλη να, να παραταθούν οι ποσοστώσεις. Είναι δύο από τα πολλά μέτρα που έχουμε εγκρίνει για να εξομαλύνουμε την κατάσταση στον γαλακτοκομικό τομέα. Και ελπίζω να διαπιστώσατε ότι πολλές από τις συστάσεις σας έχουν καλυφθεί ήδη είτε με τη μορφή στοιχείων που υπάρχουν ε, ήδη στις νέες μας προτάσεις είτε με την ε, μορφή στοιχείων που υπάρχουν στα ψηφίσματα. Έχουμε, δημιουργήσαμε κατά σύστασή σας την ομάδα υψηλού Ελπίζουμε ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2010 θα έχουμε τα οριστικά πορίσματα. Η κατάσταση είναι θετικότερη. Οι τιμές αυξάνονται, δεν υπάρχει αγορά από την παρέμβαση, διότι οι δύο τιμές είναι σχεδόν ταυτόσιμες. Τιμή αγοράς δηλαδή και τιμή παρέμβασης. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 186, είναι μια εφιστάμενη διάταξη για πολλά προϊόντα, αλλά όχι για το γάλα μέχρι τώρα. Ε, η διακύμανση των τιμών που ξεκίνησε το 2007 καταδεικνύει ότι θα πρέπει και το γάλα να συμπεριληφθεί στο άρθρο αυτό, το 186. Γιατί έτσι θα έχει τη δυνατότητα η Κομισιόν να αναλαμβάνει ταχύτερα δράση. Χθε στο, Υπουργείο, στο Συμβούλιο των Υπουργών ανήγγυλα ότι εκταμιεύουμε 280 εκατομμύρια ευρώ ενίσχυση προς τους ε, γαλακτοπαραγωγούς. Και για να γίνει αυτό ταχαίως χρειαζόμαστε νομική βάση, δηλαδή το άρθρο 186. Θέλουμε να δώσουμε τα χρήματα αυτά σε εθνικές, ε, με τη μορφή εθνικών φακέλων Κάτι το οποίο σημαίνει ότι εντάσσονται στο πλαφόν, στο ανώτατο όριο δηλαδή, των εθνικών ποσοστώσεων. Βεβαίως θα πρέπει να αποφύγουμε διακριτικές μεταχειρήσεις και να ευνοηθούν, να δοθούν αυτά τα χρήματα κατά προτεραιότητα δηλαδή σε αυτούς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Είπα ότι θα συμπληρωθεί το γάλα στο άρθρο 186 και ανήγγειλα την ε, δυνατότητα αυτή χθες ε, όταν το είπα αυτό, θα πρέπει βεβαίως να έχετε κατά νου ότι οι δημοσιονομικές αρχές, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, ε, θα πρέπει να αποφασίσουν στις 19 Νοεμβρίου να απελευθερώσουν, να δώσουν το πράσινο φως για την εκταμίεση αυτού του ποσού. Άλλα χρήματα δεν έχω να δώσω Με την εξαίρεση βεβαίω των 300 εκατομμυρίων που θα πρέπει να εκμεταμιευθούν για λόγους δημοσιονομική πειθαρχία. Το άρθρο 186, και πρέπει να το τονίσω αυτό εδώ ενώπιον σας, δεν είναι λευκή επιταγή. Στο παρόν στάδιο, η ιδιωτική αποθεματοποίηση για διάφορα προϊόντα, όπως και το τυρί, είναι μια υποψήφια λύση, αρκεί η κατάσταση στην αγορά να είναι τέτοια που να το δικαιολογεί. Το δεύτερο τμήμα της προτάσεως είναι η διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων. Υπάρχει ήδη δυνατότητα να αγοραστούν ποσοστώσεις από άλλο κράτος μέλος. Εδώ όμως προτείνουμε να μειώσουν τη συνολική τους χρήση, δηλαδή το εθνικό τους πλαφόν για τις ποσοστώσεις. Και αυτό σε θελούσια, σε θελοντική μάλλον βάση. Διότι είμαστε πεπισμένοι ότι υποχρεωτικά μέτρα δεν λειτουργούν. Κυρίως από πολιτικής απόψεως. Αυτά από την πλευρά μου και ε, είμαι στη θέση σας για να ακούσω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για το ΕΛΚ για 1,5 λεπτό ο κύριος Ντες. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο εγκρίθηκε αυτή η κατεπίγουσα, ε, το κατεπήγον αίτημα και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία. Εμείς λοιπόν δεν ε, θελήσαμε να απεκδηθούμε των ευθυνών μας. Σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους από άλλες πολιτικές ομάδες, εμείς ε, το αίτημα αυτό το θεωρούμε αιτιολογημένο σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Βεβαίω είναι αλήθεια ότι το αίτημα αυτό ε, προέρχεται καθυστερημένα από την Επιτροπή και δεν ε, είναι στο ύψος των περιστάσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει καλύτερα από το τίποτα κράτη-μέλη και οι πολιτικές ομάδες ε, έχουν προτείνει ένα πρόγραμμα το οποίο μου πρέπει να είναι δεσμευτικό για να είναι και αποτελεσματικό. Εγώ λοιπόν τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξει πλειοψηφία από αυτού και επιπλέον η δράση αυτή δεν είναι αποδεκτή για ορισμένα κράτη-μέλη γιατί ε, σε τελική ανάλυση μοιάζει με ισοπαίδωση και η επισήμανση ότι ή να δοθούν κάποιες υψηλότερες επιδοτήσεις σε κάποιες ομάδες, αυτό ε, δεν αιτιολογείται. Στο άρθρο 186 ε, θα μπορούσε κανείς να προβλέψει ειδικά μέτρα για την περίπτωση της διαταραξής της αγοράς. Εγώ όμως θα ήθελα να πω ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να περιστούν σε δύο χρόνια και αν αποδειχθούν σωστά τότε πράγματι να συμφωνήσουμε να παραταθούν. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τα 280 εκατομμύρια ευρώ. Κυρία Επίτροπε, νομίζω ότι ικανοποίησατε σε μεγάλο βαθμό ε, τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου. Ξέρω ότι δεν έχετε πια άλλα χρήματα. Παρακαλώ λοιπόν την Πέμπτη ή δυνατόν να δεχθείτε την τροποποιημένη μας αίτηση. Τροπολογία. Για για δύο λεπτά, συγγνώμη ο κύριος Ντεκάστρο signor presidente signora commissaria onorevoli colleghi innanzitutto colgo Αγαπητοί συναδελφοί, πρώτα απ' όλα δράτω με τι για να εκφράσω την πλήρη μου ικανοποίηση για το αίσθημα ευθύνης που κατέδειξε αυτή η, αυτός ο οίκος εγκρίνοντας, δίνοντας το πράσινο φως στην επίγουσα διαδικασία για να ενταχθεί το γάλα, όπως και άλλα προϊόντα, στο άρθρο 186. Οι κανόνες που ρυθμίζουν την παρέμβαση στην αγορά μας δίνουν την δυνατότητα να αποκριθούμε άμεσα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή που αφορά το σύνολο της γεωργίας και ακόμα πιο ιδιαίτερα τον γαλακτοκομικό τομέα. Και ελπίζουμε, αλλά και αναμένουμε, όπως μας είπε μόλις τώρα η Επίτροπος Φίσερμπολ, να ακούσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μέχρι τώρα αποδείχτηκαν ανεπαρκή εν ώψη της ε, βαρύτητος της κρίσεως. Η ε, ε, σημερινή το σημερινό άνοιγμα που κάνουμε βεβαίως δεν είναι λευκή επιταγή. Είναι μια κίνηση ευθύνης και υπευθυνότητας έναντι αυτής της εξαιρετικά βαρίας και οξίας κρίσης. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θέλει να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για να διασφαλίσει το δημοκρατικό έλεγχο του μέτρου αυτού και για να γίνει κάτι τέτοιο θεωρούμε ότι εκ των προτέρων θα πρέπει να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο για το πώς συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει αυτά τα νέα προνόμια, αυτές τις νέες αρμοδιότητες που τις δίδει το άρθρο 186 και με τη συμπερίληψη του Γάλακτο σε αυτό. Ευχαριστώ. Δημοκράτες και φιλελεύθεροι, 1,5 λεπτό ο κύριος Λάιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο που ήρθε εδώ για να μας εξηγήσει για το 186. Σας ευχαριστώ που απαντήσατε θετικά στα αυτό που αποφασίσαμε στις 27 Σεπτεμβρίου και που προσπαθείτε να σταθεροποιήσετε αυτή την κατάσταση σχετικά με τον γαλακτικό κομικό τομέα και για τα 280 εκατομμύρια για την αναδιάρθρωση σχετικά με το πρώτο μέρος της πρότασής σας, το, το, η ερώτηση που θέτουμε όλοι σήμερα είναι γιατί α, ε, σε αυτό το α, ε, καθυστερημένο στάδιο ε, μας ζητάτε να ψηφίσουμε αυτές τα κατυπέγοντα μέτρα ενώ έχουμε τα πρώτα θετικά σημάδια, τα πράσινα βλαστάρια αυτών των μέτρων. Όσον αφορά την πρόταση για, το, να περιλάβουμε περισσότερα προϊόντα στο 186. Νομίζω ότι οι Υπουργοί, οι Επίτροποι έρχονται στο Κοινοβούλιο ζητώντας το πράσινο φως για να λάβουν μέτρα για να λύσουν ένα θέμα. Ε, σήμερα να μας ζητάτε να δώσουμε αρμοδιότητες εξουσίες στην Επιτροπή ε, για να δουν ε, τι μέτρα θα πρέπει να λάβουν. Από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτά που είπατε προηγουμένως αναφέρατε, ότι χρειάζεστε αυτές τις επιπλέον αρμοδιότητες για τα 280 εκατομμύρια. Έτσι είναι. Γι' αυτό απαιτείτε αυτές τις επιπλέον εξουσίες και αρμοδιότητες. Ε, ε, ίσως μπορεί, δεν ξέρω αν αυτό είναι μια λευκή επιταγή που δίνουμε στην Επιτροπή. Είπατε ότι ότι αν έχετε άλλες ιδέες μέτρων που μπορούν να ληφθούν, ίσως δεν έχει αυτό οικονομική σημασία. Θα δώσουμε αυτές τις αρμοδιότητες αν είναι περιορισμένες και αν εφαρμόζονται μόνο σε έκτατες περιστάσεις. Για τους πράσινους, 1,5 λεπτό ο κύριος Χάσλινγκ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτέλους λοιπόν βλέπω κάτι να γίνεται. Υπάρχει κίνηση στη συζήτηση. Η Επιτροπή τώρα Καλύτερα να αναλάβει πλήρω την ευθύνη. Σήμερα το πρωί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα θέλαμε να συμπεριληφθεί περισσότερο το Κοινοβούλιο. Και για να είμαστε απόλυτα σαφεί, εμεί δεν είμαστε κατά των οικονομικών ενισχύσεων. Πρέπει όμω να είναι σαφέ ότι πρόκειται για σταγόνα στον ωκεανό. Κυριολεκτικά σταγόνα στον ωκεανό. Και οι αποφάσει του Λουξεμβουργού δυστυχώ δεν συνέβαλαν στο να ρυθμιστεί η ζήτηση και η προσφορά. Κάτι που είναι πραγματικά καθοριστικό. Ε, ναι, συμφωνούμε με τις ε, εθελοντικές αγορές ποσοστώσεων, αλλά αυτό δεν θα έχει καμία σημαντική αποτελεσματικότητα. Το είπαμε ήδη. Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και να εφαρμόσουμε μια μακροπρόθεσμη πολιτική. Και να δούμε τι μας είπε το ελεγκτικό συνέδριο. Μας είπε λοιπόν ότι στο μέλλον πρέπει να ρυθμίζουμε την προσφορά, αλλιώς το σύστημα δεν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Και χρειαζόμαστε ποιοτικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τέτοια πολιτική γάλακτος. Νομίζω λοιπόν ότι το συντομότερο δυνατόν πρέπει να απομακρυνθούμε από τις επιδοτήσεις εξαγωγών γιατί προηγουμένως ήδη κάποιοι επισήμαναν ότι είχαν ολέθριες συνέπειες. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια επίκαιρη πολιτική που να αντιμετωπίζει και την κρίση και περιμένουμε και κάποιες απαντήσεις από την Κομισιόν για το μέλλον. Δυστυχώς μέχρι τώρα η Κομισιόν δεν μας έδωσε τις απαντήσει επενδύσεις αυτές. Ε, ε, μας ε, χρειάζονται όμως για να βοηθήσουμε τις οργανώσεις παραγωγών και για να μπορούν και αυτοί να επιβάλλουν κάποιες δικές τους απόψεις στις αλυσίδες καταστημάτων. Για τους συντηρητικούς και μεταθυμιστές, ένα λεπτό ο κύριος Νίκολσον. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω αυτήν την απόφαση ε, εχθές ε, στην Επιτροπή και σήμερα ε, νομίζω ότι έχουμε πλέον τη δυνατότητα να επιφέρουμε φως, περισσότερο φως στην κατάσταση. Η απογοήτευση που νιώθουν πολλοί γαλακτοπαραγωγοί είναι ότι, όπως είπε ο κύριος Λάιον, ε, είδαν να υπάρχουν ε, κάποιοι σπόροι που θα ευδοκιμήσουν στο μέλλον, όμως δεν έχουν δει ακόμα τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ε, νιώθουν λοιπόν απογοητευμένοι γιατί πολλοί για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν υπό ασφικτική οικονομική πίεση. Πάντως, κυρία Επίτροπε, καλό είναι αυτό που το συζητάμε, γιατί τώρα Τώρα πλέον όλοι δεχόμαστε ότι πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 186 έτσι ώστε να ενισχύσουμε τους παραγωγούς των στομότων δυνατών. Ε, καλή ήταν αυτή η ιδέα που υποβλήθηκε για την τροπολογία. Εγώ θα στηρίξω την ε, τροπολογία αυτή για τα δύο ή τρία χρόνια που προβλέπει. Ε, βέβαια, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τον τομέα. Ευχαριστούμε. Για την Γκουε. Δύο λεπτά ο κύριος Λεγιαρικ. Γιαρικ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω σήμερα το βράδυ ότι οι διατάξεις, οι χρηματικές που προτείνεται είναι μια σταγόνα μέσα στον ωκεανό της απόγνωσης που ζουν σήμερα οι αγρότες. Θα ξεμπλοκάρετε 280 εκατομμύρια ευρώ ενώ πριν μερικές εβδομάδες είχε γίνει λόγος για 600 εκατομμύρια. Θα δώσετε μια φορά λοιπόν 1000 ευρώ σε αγρότες που σήμερα χάνουν από 100 έως 200 ευρώ την ημέρα. Ζητούμε, ζητούμε λοιπόν ένα πραγματικό κατεπήγον πρόγραμμα και όχι ένα τσιρότο για να θεραπεύσει κανείς έναν καρκίνο. Δεν θέλετε για ένα μεγάλο πρόγραμμα ε, για την σφαγή ε, αγελάδων και κλείσιμο αγροκτημάτων. Ε, γιατί έτσι θα, θα καταστρέψετε το μέλλον της γεωργίας των νέων γεωργών, αυτοί που παράγουν τυριά ποιότητας και διαφυλάσσουν το περιβάλλον περιβάλλον. Πώς να το προτείνετε αυτό όταν τόσες οικογένειες στην Ευρώπη δεν έχουν πρόσβαση στα τρόφιμα αρχίζοντας από το γάλα. Αύριο με το πρόγραμμά σας θα έχουμε έλλειψη γάλακτος. Τη στιγμή όπου τόσο επενούν το συνθήκη της Λισαβόνας εκπλησόμεθα που θέλετε να εφαρμόσετε αυτό το άρθρο 186 του κανονισμού που θα σας δώσει πλήρες εξουσίες. Τις πλήρες εξουσίες τις είχατε και το γεγονός ότι είχατε αυτές τις απόλυτες εξουσίες σας έκανα αποφασίσετε την απελευθέρωση των ποσοστώσεων που μας βήθησε στην κρίση που γνωρίζουμε σήμερα και ευνοεί μόνο τους εμπόρους και τους βιομηχάνους. Σήμερα ε, το ελεγκτικό συνέδριο δείχνει ότι από το 2000 έως το 2007 οι τιμές κατανόλωσης των απογαλακτοκομικών αυξήθηκαν 10% ενώ οι τιμές για τους παραγωγούς μειώθηκαν κατά 6%. Κύριε Επίτροπε, άλλη μια φορά σας λέω ότι είναι κατεπήγον, πολύ κατεπήγον να βοηθήσετε μαζικά την γεωργική εργασία με ένα μεγάλο ταμείο επίγον ε, και να επανέρθετε σε ελάχιστες τιμές και να μην αφήσετε την καπιταλιστική αγορά να καταστρέψει τους αχρότες μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Το λόγο έχει για τους μη εγγεγραμμένους για 1,5 λεπτό η κυρία Μορβάη biztos ότι, természetesen igennel ξέρω ότι αυτό που προτείνεται δεν θα λύσει την κατάσταση για τους αγρότες. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση για σας. Τι δίδαγμα πρέπει να αντλήσουμε από αυτή την κρίση. Έχετε εξαγάγει κανένα συμπέρασμα από αυτή την κρίση. Κυρία Επίτροπε, ε, δεν ε, είναι η συνέπεια αποφάσεων, κακών αποφάσεων αυτή η κατάσταση και είναι η συνέπεια μιας αγροτικής πολιτικής που είναι μια αποτυχία. Τι θα υποσχεθείτε για το μέλλον ε, στους γεωργούς. Πώς θα αποφύγουν παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον. Αυτή είναι η ερώτηση που σας θέτω για να έχω μια λεπτομερή απάντηση στην πρώτη αυτή ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση, είπατε χθε ε, στην ακρόαση της Επιτροπής ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν αυτά τα ποσά. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα κράτη-μέλη μπορούν με δίκαιο τρόπο να κατανείμουν τα χρήματα αυτά ούτως ώστε να μην είναι ε, οι αγροτροφικές μονάδες οι μεγάλες, ε, τα μεγάλα εργοστάσια που θα ευνοηθούν αλλά οι μικροί που έχουν περισσότερη ανάγκη και που εξαρτώνται από τη βοήθεια αυτή για την επιβίωσή τους και κυρίως αυτοί που βρίσκονται στην δυσκολότερη κατάσταση αλλά κυρίως οι μικροί αγρότες των νέων κρατών μελών. Πώς θέλετε να θέσετε τέρμα σε αυτήν την ε, απαράδεκτη διάκριση που σημαίνει για μας τους Ούγγρους παραμπτός χάρη χρειάστηκε να ανοίξουμε 100 τις, 100 τις αγορές μας για την υπόλοιπη ένωση και ως αντάλλαγμα λάβω ένα μικρό κλάσμα της αγοράς. Πώς θέλετε να θέσετε τέρμα σε αυτήν την ανισότητα. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Λαβία. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, εκτιμώ την στάση της Επιτρόπου που ήλθε στο Στρασβούργο για να μας ε, εξηγήσει την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των παρεμβάσεων που προτείνονται, παρόλο που είναι ανεπαρκή η περιγραφή των λεπτομεριών, θεωρώ ότι αποτελεί μια θετική άγουσα για την επίλυση των προβλημάτων που ζουν οι εκτροφείς. Δεν νομίζω όμως ότι αυτές οι επιβάσεις από μόνες τους μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπερψηφίσουμε την ε, πρόταση τροποποίησης των άρθρων 78-79 για το, το, του κανονισμού 2034. Στο άρθρο 78, στα στοιχεία α και β, προβλέπεται ε, διαφορετική προστασία διαφορετικών προϊόντων. Ε, ενώ ε, για άλλα προϊόντα ας πούμε χειριοκρέας και ελαιόλαδο ή ελιές υπάρχει άλλη αντιμετώπιση αυτή είναι μια ανακολουθία ε, καταδικαστέα στο όνομα του ΕΛΚ ε, προτίθεμαι να υποβάλω μια τροπολογία σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιοδήποτε δράση δυνάμει του άρθρου 186. Αυτή η τροπολογία μπορεί να συνδυαστεί και, μια σχετική, και με μια σχετική των σοσιαλιστών τροπολογία. Θα ήθελα επίσης και τέλος, όπως έκανα και για το ψήφισμα της 17ης Σεπτεμβρίου, να ζητήσω από την Επιτροπή την αύξηση των ντεμίνιμις για όλα αυτά τα προϊόντα, ανεξάρτητα από τα εθνικά πλαφόντα που υπάρχουν για το συγκεκριμένο προϊόν. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Λαβία. Για ένα λεπτό κύριο Καπούλα Σάντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, όλοι δυστυχώ γνωρίζουμε την οξύτατη κρίση που πλήττει τον γαλακτοκομικό τομέα στην Ευρώπη. Η πολιτική μου ομάδα έχει πολλά και ζητήσει επίγοντα μέτρα για να σώσει από την καταστροφή τις χιλιάδες των αγροτών και των εκτροφέων που απειλούνται από αυτήν. Γι' αυτό υποστηρίξαμε αυτήν την παρέμβαση και γι' αυτό υποστηρίξαμε και παρέμβαση άλλων πολιτικών ομάδων που είχαν το ίδιο στόχο. Γι' αυτό δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω την πρωτοβουλία της Κομισιόν, έστω και αν μας φαίνεται εντελώς ανεπαρκής. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η σοσιαλιστική ομάδα ε, πρότεινε και το την τροπολογία αυτή. Γι' αυτό υπερψήφισε το ψήφισμα και θα συνεχίσουμε να ζητούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται διαρκώ για τις αρμοδιότητε που χωρούμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και τα μέτρα που θα ανάλευε δυνάμει του άρθρου 186. θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα, ούτω ώστε να επανεξισορροπήσουμε την αγορά για να έχουν ένα αξιοπρεπέ εισόδημα οι γεωργοί μας. Εξάλλου, αυτός είναι ο στόχο και τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από ό,τι μα είπε η κυρία Επίτροπος. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, η κυρία Πόλσεν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, βεβαίως ε, είναι απολύτως απαραίτητο να αντιδράσουμε ταχύτατα και αυτό πάντα όταν εμφανίζονται κρίσεις σε διάφορες τομείς. Ε, αυτό το βιώσαμε στις ε, τράπεζες, στο βιομηχανικό τομέα, αλλά και στους γεωργούς. Πρέπει να πούμε, οι κρίσεις αυτές θα υπάρχουν, θα υπάρχουν πάντα. Την επόμενη φορά, ίσως να μην είναι το γάλα, να είναι τα σιτηρά ή κάποιο άλλο προϊόν. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω κάτι που αφορά την ουσία της συζήτησης. Δηλαδή, όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν μπορούμε πάντα να λύνουμε τα οξέα προβλήματα. Και οφείλουμε να έχουμε το θάρρος και να επιδεικνύουμε πολιτικό προγραμματισμό έτσι ώστε να ε, χαράξουμε μια κοινή γεωργική πολιτική η οποία θα είναι διάρκειας, ευέλικτη, μια πολιτική η οποία θα αντιμετωπίζει τις ε, ολέθριες συνέπειες που απορρέουν από την αστάθεια των τιμών. Εγώ λοιπόν εύχομαι να υπάρχουν ζωντανές ε, κοινότητες γεωργών, αλλά υπάρχουν αυτές, πρέπει να υπάρχουν και γεωργοί και ζώα. Ευχαριστώ κύριε Πόλσεν. Δεν βλέπω τον κύριο Μποβέ στο έδρανό του. Είναι εδώ ο κύριος Μποβέ. Äh, äh, Κοιτάξτε, η κυρία Ζήμποβε δεν μπορούσε να είναι εδώ, γι' αυτό πήρα εγώ και πάλι το λόγο. Και έχω να κάνω κάποιε ερωτήσει προ την κυρία Επίτροπο. Ε, κατά πόσον πραγματικά πιστεύει ότι θα ε, εξουδετερωθούν πλέον οι διαμαρτυρίες με τα κονδύλια που θα καταβληθούν. Σήμερα το πρωί είπα ότι αυτή την απόφαση του Κοινοβουλίου την θεωρώ λευκή επιταγή και δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Κομισιόν. Είπα ότι η Κομισιόν κατά την άποψή μου δεν είναι τμήμα της λύσης αλλά τμήμα του προβλήματος και επιμένω επ' αυτού. Βεβαίω ε, πρέπει κανείς ε, να βλέπει την αλήθεια κατάματα. Ε, δεν παραβλέπω το τι αποφασίστηκε σήμερα το πρωί. Θέλω να πω στου συναδέλφου ότι οφείλουμε να περιορίσουμε την ισχύ των μέτρων σε ένα προβλέψιμο χρονικό διάστημα έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί και πάλι να αναλάβει τα ενία. Πάντως κυρία Επίτροπε θέλω να κάνω μια ερώτηση πρέπει να συνεχίσουμε να προάγουμε την αναδιάρθρωση. Είπατε εσείς. Και τι εννοείται αναδιάρθρωση. Θεωρείτε ότι είναι σωστό να εξακολουθήσουμε να εκταμιεύουμε κονδύλια έτσι ώστε να κλείσουν μικρές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να παραδοθούν σε μεγαλύτερες. Αυτή η πολιτική δεν οδηγεί πουθενά. Οφείλουμε λοιπόν να ε, δούμε τις δομές ε, στις μειονεκτούσες περιοχές, εκεί να διοχετεύσουμε στοχευμένα τα κονδύλια έτσι ώστε να διατηρηθούν εν ζωή οι αγροτικές αυτές εκμεταλλεύσεις που κινδυνεύουν. Κύριε ευχαριστώ και τώρα. Ο κύριος Βλόσοβιτς, ούτε αυτός όμως βλέπω είναι στο τρανό Πού έχει κρυφτεί πουθενά. Καλά. Πάμε τότε στον επόμενο. Φερέιρα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αποτυχία της πολιτικής μας για τον γαλακτοκομικό τομέα. Παρ' όλα αυτά διατηρεί τον ίδιο προσανατολισμό. Τα εκατομμύρια που αναφέρατε υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών που έχουν ε, οι παραγωγοί. Αντίθετα αυτό που μας λέτε πρέπει να προχωρήσουμε προς μία ΚΑΠ ε, που θα, δεν θα, ε, που θα ε, αν συνεχίσουμε δηλαδή αυτήν την στρατηγική θα καταστρέψουμε όλη την ΚΑΠ. Θα χάσουμε δισεκατομμύρια και οι γεωργοί θα εγκαταλείψουν ε, ε, την αγροτική τους δραστηριότητα. Θα περιμωθεί η ύπεθρος με καταστροφικούς κοινωνικούς και οικονομικούς αντικτύπους. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια μεγαλύτερη παρέμβαση, με μεγαλύτερα μέσα από όσα κοινοποίησατε τώρα. Και βεβαίως πάνω απ' όλα πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε μέτρα μεγαλύτερου, ευρύτερου βεληνικούς, όχι μόνο πολιτικά ή συγκεκριμένα όπως μία ετήσια αύξηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Θα πρέπει να σταματήσει και βεβαίως ε, η ανάκληση της απόφασης να σταματήσει το σύστημα των ποσοστώσεων. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Ντότζ. Thank um, όπως οι περισσότεροι βουλευτές εδώ και εγώ σήμερα θέλω να ταχθώ υπέρ της πηγούς διαδικασίας του 186. Οποιαδήποτε ενίσχυση είναι επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση του κλάδου αυτού, ιδίω όσον αφορά το πώ θα επιβιώσουν οι μικρέ οικογενειακέ εκμεταλλεύσει, όπω είναι η κατάσταση στην Βόρεια Ιρλανδία. Χρειάζονται επομένω να επιφέρουν κάποιε μεταλλαγέ στο 186, ούτω ώστε να μπορέσουν τα, τα 280 εκατομμύρια να εκταμιευτούν. Εάν το κάνετε αυτό, τότε έχετε την υποστήριξή μα και ελπίζουμε ότι θα εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα, θα πληρωθούν, θα διανεμηθούν ταχύω, διότι οι περισσότεροι των γεωργών έχουν περιμένει πάρα πολύ, ούτω ώστε να μπορέσουν να λάβουν τα προβλεπόμενα. Και δεν σα πω, έχω την ότι έχω εκπλαγεί από αυτά που προβλέπονται στι διατάξει 65 με 84 τη προτάσει σα, διότι είναι σίγουρο ότι αυτά δεν μπορούν να έχουν καμία επίπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αναδύονται ένα σωρό ερωτηματικά σχετικά. Ιδίω εκεί που λέει ότι, ότι, ότι θα, θα, θα, έχουμε κάποιο είδου ε, ανισότητα στον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών, κάτι που έρχεται τη κατάφραση με την ισχύουσα πολιτική. Ευχαριστούμε κύριε Δόζλιο Πρόεδρο. Και τώρα για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριο. la palabra por Ενάμιση λεπτό συμπαθάτε με, λέει ο Πρόεδρος. Μπεσί. Merci, Monsieur Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χρειάζεται να υπάρχει συνέπεια στην πολιτική. Και ε, εδώ, όπως είμαστε τελευταία εβδομάδα, πάρα πολλοί από εμά ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρα, μέτρα άπαξ και τώρα ήρθε η ώρα των απαντήσεων, εμείς θα τις ψηφίσουμε. Όμως ε, συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε, ότι πάρα πολύ αργά, γιατί είπατε πολλές φορές με το, με το τσιγκέρι, της βγάλεις σε σχέση με αυτά που εμείς πρεσβεύαμε, σε σχέση με αυτά που είπε το Συμβούλιο. Οπότε αυτό το ποσό δεν επαρκεί, το οποίο πρόκειται να εκδεμευτεί ε, για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες, γιατί πολλοί είπαν τι θα γίνει μακροπρόθεσμα όσον αφορά τα προγράμματα, αφορά τις ποσοστώσεις, τι θα γίνει, δυνατόν κανένας να έχει ε, μέτρα κανονιστικά και μέτρα διαχείρισης θα πρέπει και τα δύο να γίνουν ούτως ώστε να μπορεί κανένας να αντιμετωπίσει αυτές τις ε, κρίσεις που σοβούν συνέχεια στον τομέα. Όμως αυτό το θέμα δεν είναι ε, που συζητάμε απόψε. Το θέμα τι θα γίνει με το 186. Έχω μια ερώτηση, κυρία Επίτροπε, μια ερώτηση απλή. Το 186 θέλετε να το επικαλεστείτε για να κάνετε τι, από πότε και με ποιο τρόπο. Ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπεσιού. Και τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Γκαρθία Πέρεθ. Εδώ και ένα μήνα θα συζητάμε εδώ για αυτό το ψήφισμα του Κοινοβουλίου αλλά και τι προτάσει σα όσον αφορά την παρέμβαση στα γαλακτοκομικά. Σήμερα έχουμε αυτά τα δύο φρέσκα μέτρα, δηλαδή το πώ θα αλλάξει η διαχείριση των αποστάσεων και το 186 είναι μέτρα τα οποία θα πρέπει να, να τα τόσο όσο γίνεται πιο γρήγορα όπω και συζητήσετε. Και όμω, κύριε Επίτροπε, χρειάζεται ο κλάδο ενό είδου ε, ε, συνολική διαχείριση. Και όχι να υπάρχουν τέτοια εμβαλωματικά μέτρα τα οποία τα συζητάμε εδώ και τόσου μήνε, διότι θέλουμε να είναι πανευρωπαϊκέ οι λύσει. Κοινού χαρακτήρα και γι' αυτό αυτό το οποίο είπατε, να υπάρχουν αυτέ οι ελάχιστε ενισχύσει και να αυξηθούν, όμω αυτό θα φέρει κάποιε τρευλώσει και αυτό πρόκειται να είναι φραγμό στη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Η τελευταία μα σκέψη είναι ότι είπατε για αυτά τα 200 380 εκατομμύρια σε ενίσχυση και βεβαίω εμεί χαιρετίζουμε αυτή την κίνηση. Όμω σα υπενθυμίζουμε κύριε Επίτροπε ότι στο κοινοβούλιο τούτο έχουμε ήδη περάσει ένα ψήφισμα που λέγαμε ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα άλλο ε, ποσό 600 εκατομμύριων τόσο ώστε να αντιμετωπίσει ο κλάδο την κρίση. Ευχαριστούμε κύριε Καρθιαπάρη και τώρα για ένα λεπτό έχετε το λόγο κυρία Ράιμερ. Αξιότιμε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σε αυτή την τροπολογία του άρθρου 78 ε, και 79 εγώ ως ε, γεωργός ε, βλέπω ότι καλά τα πάτε ως προς την γεωργική μεταρρύθμιση και αυτό θα ωφελήσει τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό προς το μέλλον. Μέχρι τώρα το σύστημα των ποσοστώσεων ήταν εις βάρος των γαλακτοπαραγωγών και κατόπιν τούτου αυτοί ήταν αναγκασμένοι να ε, κυνηγάνε τις εξελίξεις. Τώρα αρχίζει κάπως να βελτιώνεται την κατάσταση. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι η Κομισιόν την έκκληση του Κοινοβουλίου για ταχύτατα μέτρα θέλει να την εκμεταλλευτεί. Και αυτό το κάνει με το ότι λίγο πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας προσπαθεί με το άρθρο 186 να εξασφαλίσει κάποιο χώρο ε, κινήσεων ανεξάρτητα από το Κοινοβούλιο. Εγώ αυτό το απορρίπτω. Θα μπορούσα όμως να δεχθώ το Κοινοβούλιο να δώσει σε περίοδους κρίσης σε κάποιο χρονικό διάστημα ελιγμών στην Κομισιόν. Και αυτό θα μπορούσε να στηριχθεί και με τροποποίηση του κανονισμού του άρθρου 142 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Ashworth. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ο γαλακτοκομικός τομέας αντιμετωπίζει προβλήματα, βρίσκεται σε κρίση. Συγχαίρω την κυρία Επίτροπο για την έγκαιρη παρέμβασή τη, σωστή αυτή. Ε, τα 280 εκατομμύρια ευρώ είναι ρεαλιστικό το ποσό και νομίζω ο τομέας ε, θα το δεχθεί με μεγάλη του χαρά. Επίσης, ε, το άρθρο 186 είναι απαραίτητο για να μπορεί κανείς να δώσει τα χρήματα αυτά έγκαιρα στους παραγωγούς και αυτό το στηρίζω. Στηρίζω παρότι θα προτιμούσα την παραχώρηση αυτή να την περιορίσουμε μέχρι το 2013 το αργότερο. Τη στηρίζω λοιπόν. Όσον αφορά τώρα ε, το σύστημα των ποσοστώσεων γνωρίζω ότι εκεί θα συμπεριληφθούν εξουσιοδοτήσεις για μια υπερβολική ενίσχυση ε, μάλλον υπερβολική πρόσφαση σε ε, παραγωγούς που ξεπερνάνε τις ποσοστώσεις, αυτό σημαίνει ότι τιμωρούμε τους νέους που είναι το μέλλον του τομέα και περνάει ένα λανθασμένο μήνυμα. Ζούμε λοιπόν σε μια πολύ ευμετάβλητη αγορά και αυτό που χρειάζεται ο τομέας δεν είναι βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις αλλά μακροπρόθεσμη στρατηγική. Εγώ για μεγάλο χρονικό διάστημα ήμουνα οπαδός της ε, Κομισιόν που είχε έτσι ένα μακρόπνο όραμα για το μέλλον και την καλό να επανέλθει σε αυτό. Τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και όχι τις βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Καλινόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ελπίζω ότι κανένας παραγωγός δεν είναι πίσω από αυτά. Η απόφαση υποστήριξης των γαλακτοπαραγωγών με 280 εκατομμύρια του χρόνου είναι καλό σημάδι. Αλλά παραμένουν ε, βασικά ερωτήματα για το από πού θα πάμε από εδώ ε, και πέρα που δεν θα έχουμε παραγωγή γάλακτος και γαλακτοπαραγωγούς στο μέλλον και το μέλλον των ποσοστώσεων για την παραγωγή γάλακτος. Υπάρχουν δύο τάσεις για την ώρα. Η πρώτη είναι αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ που βαθμία αυξάνει της αναθεώρησης της ΚΑΠ που οδηγεί βαθμία στην κατάργηση των ποσοστώσεων το 2015 και δεύτερον στη μείωση, τάση της μείωσης της προσφοράς γάλακτος και οι δύο τάσεις αυτές είναι αντιφατικές. Είμαι υπέρ της διατήρησης των ποσοστώσεων, αλλά εάν ε, έχει κάποιο, ε, ε, η κατανομή γίνεται με κριτήρια δίκαια μεταξύ των κρατών μελών. Είναι δύσκολο να υπάρχουν δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια, αλλά αξίζει να προσπαθήσει κανείς όσον αφορά την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 186 βεβαίως, αλλά πρέπει να υπάρξει ένας ορισμός του ρόλου και των μέσων που θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Καλινάφσκι. Τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, αν ε, ξεχάσουμε ε, ότι η κρίση αυτή άρχισε από το μηδέν ε, και πριν από αρκετούς μήνες είπατε ότι θα αυξηθούν σημαντικά οι τιμές γάλακτος ενώ μειώθηκαν κατά το ίμιση σε, σε πολλά κράτη-μέλη και νομίζω ότι η πρόταση είναι θετική από αυτήν την άποψη. Στην δική μου εκλογική περιφέρεια έχουμε μικρούς, μικρές εκμεταλλεύσεις και μεσές που επιβιώνουν ε, ή ε, ίσα ίσα ή βρίσκονται δίπλα στην πτώχευση. Έχουν λοιπόν μεγάλες δυσκολίες ε, και η στήριξη των, των τραπεζών δεν ωφελεί. Κύριε Κέλλη, σας παρακαλώ να μιλάτε λίγο πιο αργά παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος. Τα 280 εκατομμυρία που αναγγέλθηκαν είναι ευπρόσδεκτο, αλλά είναι κάτι το μικρό σχετικά με το ευρύ πρόβλημα. Ε, το Σεπτέμβριο είπαμε ότι έπρεπε να ψηφιστούν 600 εκατομμύρια για να ε, επιδείξουμε αλληλεγγύη στους μικρούς ε, αγρότες. Πρέπει να διατηρηθεί αυτό το κονδύλι και μετά θα πρέπει η Επιτροπή να ασχοληθεί με όλο το θέμα της προσφοράς γάλακτος. Μέχρι ότου καλυφθεί αυτό θα έχουμε περισσότερα προβλήματα και θα έχουμε και πάλι τις, τις ίδιες κρίσεις. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Δίνω το, την, στην ε, κυρία Γέγκελ για ένα λεπτό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ναι, πρέπει να συμφωνήσουμε το γάλα να συμπεριληφθεί στο 186. Και ελπίζω να το πράξουμε αυτό αύριο. Δεν μπορούμε συνεχώς ε, να ασκούμε κριτική στην Κομισιόν, ότι καθυστερεί, ότι μας κυνηγά από πίσω ε, και ξαφνικά έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει ταχύτητα. Πρέπει λοιπόν να της την προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα και βεβαίω ε, με την βούλησή μας να ασκούμε έλεγχο τα 280 εκατομμύρια ευρώ. Τα έφυξαν πάρα πολύ πράγματι σταγόνα στον ωκεανό. Όμω πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και τώρα βρισκόμαστε στο τέλο του προπολογισμού. Ε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον χρήματα. Ε, τι θα κάνουμε λοιπόν εν ώψη αυτή τη κατάσταση. Εμείς επιθυμούμε αυτά τα 280 εκατομμύρια να τα λάβουν εκείνοι οι παραγωγοί που έχουν θυγεί βαρύτατα από την κρίση. Μιλάμε για αγορά, αλλά πρόκειται για ανθρώπου για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που σε άλλες περιπτώσεις λέμε όλους αυτούς θέλουμε να τους προστατεύσουμε. Κυρία Επίτροπε, εσείς στηρίζετε το ε, Ταμείο Γάλακτος. Σήμερα ο συνάδελφός σας που μίλησε το στήριξε, χάρηκα πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτό το μήνυμα και αυτά τα κονδύλια περιλαμβάνονται στον προπολογισμό του 2010. Ευχαριστώ στο, στο, στο κομμάτι του Κατζηδία και έχει, για να δευτώ, η κυρία. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, και εγώ υπερψήφισα την επίγουσα διαδικασία γιατί θεωρώ ότι η ενσωμάτωση του γάλακτος 186 ήταν επίγον θέμα το έπρεπε να ασχοληθούμε με αυτό επίγοντος τόσο για οικονομικούς όσο και για κοινωνικούς λόγους. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα, την Πορτογαλία και μια περιοχή, τις Αζόρες, όπου ο γαλακτοκομικός τομέας έχει τεράστια σημασία διότι ε, ε, η σχετική δραστηριότητα γίνεται σε εύθραυστο κοινωνικό περιβάλλον και ιστό. Πρέπει να διατηρηθούν οι μετά το 2015. Τα προτινόμενα μέτρα είναι ανεπαρκή, μεν απαραίτητα και επίγοντα δε. Με ανησυχεί επίσης το νέο πακέτο των υπήν αρμοδιοτήτων που δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι ε, έχει αποδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα στη στιγμή αυτή της κρίσης, ότι καθυστερεί και να λαμβάνει πρωτοβουλίες και δεν έχει το απαραίτητο πολιτικό θάρρος. Ναι λοιπόν στο 186, ναι στη συμπερίληψη του γάλακτος στο 186, αλλά όχι λευκή επιταγή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κυρία Πατράο. Για ένα λεπτό η κυρία Γιάρ. Perdón, el señor... Συγγνώμη, λέει ο ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, κυρία Επίτροπε, να στηρίξω καταρχήν το έτοιμά σας, αλλά να ασκήσω κριτική σε ένα θέμα, στο εθελοντικό πρόγραμμα επαναγοράς των ποσοστώσεων. Ε, τελικά αν ένα τέτοιο πρόγραμμα ε, στεφθεί από επιτυχία αυτό μπορεί να γίνει μόνο δεσμευτικά και όχι προαιρετικά. Αυτή την ε, προαιρετική δυνατότητα επαναγοράς ποσοστώσεων τη βρίσκω αντιπαραγωγική και ενδέχεται να αναγκαστούμε να αναζητήσουμε κάποια λύση για τις ε, ποσοστώσεις και όχι μόνο αυτό, αλλά θα επιδεινώσουμε και τις ε, δυνατότητες ε, εξυγίανσης. Εγώ τα απορρίπτω όλα αυτά, κυρίως διότι πάβει σιγά σιγά να ισχύει το μέτρο των ποσοστώσεων. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν κάποια εξισορρόπηση για να αντιδράσει μόνη της η αγορά. Για αυτούς τους ε, λόγους ε, θα καταψηφίσω αυτό το κομμάτι της πρώτης Κομισιόν. Θα υπερψηφίσω όμως την πρόταση στο σύνολό της. Ο κύριος Κορτές έχει το λόγο. Κορτές. Κορτές. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, όντως πρόκειται να ληφθούν κάποια μέτρα τα οποία θα κατευθύνονται ή στο να υπάρξει μια εν μέρη λύση του προβλήματος των γαλακτοκομικών. Ξέρουμε όλοι πώς έχει κατάσταση με τις ε, εκμεταλλεύσεις των ε, γεωργών μας και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα μέτρα για αυτούς και τις οικογένειές τους διότι οι αγρότε μας δεν θέλουν βέβαια να ζουν ε, από επι, επιδοτήσεις, ζητούν όλοι να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να μπορούν να έχουν κάποια αξιοπρεπή, δίκαιη εύλογη τιμή για το προϊόν τους και αν μπορούν να βρούμε σε επενδύσεις. Οπότε και αυτόν τον τρόπο εμείς σας υποστηρίζουμε, δείχνουμε εμπιστοσύνη ε, και, στους, ε, και σε εσάς και στους ε, γεωργούς μας, τους κτηνοτρόφους. Οπότε θα πρέπει να, να ταινίσουμε τις καινούργιες μεταρρυθμίσεις που θα ζητούν εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρε και δίνω λόγο στην κυρία Μακ Γκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα πιο σημαντικά που ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ότι οι τιμέ αγορά έχουν αρχίσει να τον ενιούσα και οπότε και εμεί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το μήνα θα περάσει στου κτηνοτρόφου. γιατί ε, βεβαίω του αρέσουν αυτά τα εκατομμύρια των ισχύσεων αλλά ε, από κάθε επιδότηση είναι πολύ πιο σημαντική κάθε δεκάρα που θα πάνε στην αγορά τιμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι πέραν των επικρίσεων να σταματήσουμε την πανέβαση να την ε, επικρινούμε διότι η πανέβαση χρησιμοποιείται και στο να στηρίζει μέσα ακόμα και σε αυτά τα τραγικά επίπεδα τα σημερινά. Επομένως είναι πάρα πολύ αυστηρές και άδικες αυτές οι επικρίσεις. Συμφωνούμε με το να γίνει επίκληση 196 αν θέλετε να εκταμιάσετε ότι αυτά τα 180 ε, εκατομμύρια θεωρώ ότι δεν είναι το σημαντικό ποσό, μάλλον συμβολικό είναι. Άρα συμπεράσματα, μαθήματα να δούμε τι θα γίνει μετά το 2013 με τη μεταρρύθμιση. Έχουμε την ομάδα ψηλοεπέδου και έχουμε κάποιε πολιτικέ ομάδε που σήμερα ε, είναι υπέρ τη ενίσχυση του τομέα. Ε, Εσεί για κοιτάξτε και τότε όταν έρθει η ώρα να υποστηρίξετε να, έχει κατάλληλη προκοδότηση μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ μετά το 2013. Αλλιώ αυτά που λέτε είναι κενά λόγια. Ευχαριστώ κύριε Μαγίνο Λεπρόδο και δίνω το λόγο στον κύριο Πόβε. Με συγχωρείτε, πρέπει να ήμουν εδώ προηγουμένω, αλλά είχα κάποια άλλη υποχρέωση. Εξηγούσα στου Γάλλου ακροατέ, τι συνέβη χθε στο Λουξεμβούργο. Νομίζω ότι η απόφαση του Συμβουλίου είναι κακή απόφαση. Κακή απόφαση διότι η μόνη λέξη που έχουμε στο κείμενο είναι αναδιάρθρωση περάσαμε από 480.000 παραγωγούς το 84 σε λιγότερο από 88.000 σήμερα. Σήμερα μας λένε ότι πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των παραγωγών και ότι τα χρήματα που θα ανακτήσουμε είναι στο κείμενο θα χρησιμεύσουν για τους παραγωγούς που ξεπέρασαν, που ηρεπερεύησαν τις ποσοστώσεις τους. Θα πρέπει ε, στις πιο δύσκολες ζώνες να μειώσουμε τον αριθμό των γαλακτοπαραγωγών. Αυτό ε, δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα χρήματα αυτά, τα 280 εκατομμύρια εκατομμύρια που προβλέφτηκαν, λέχθηκε ήδη, είναι 50 ευρώ ανά εκμετάλλευση ε, το μήνα για ένα χρόνο. Είναι μια σταγόνα, μια σταγόνα, είναι περιφρόνηση σε σχέση με την κρίση που ζουν οι αγρότες. Σχετικά με το άρθρο 186 νομίζω ότι σε μια στιγμή όπου θα έχουμε την συναπόφαση για το θέμα της γεωργίας είναι απαράδεκτο να ξαναδώσουμε λευκή επιταγή απόλυτη εξουσία στην Επιτροπή. Μία ένα λεπτό, ο κύριος Νικουλέσκου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την Επίτροπο, την οποία ευχαριστώ για την παρουσία της εδώ. Τα ποσά που υποσχέθηκαν για τον γαλακτοκομικό τομέα θα δοθούν στα κράτη-μέλη βάσει ιστορικών λόγων και τα ορισμένα κράτη-μέλη δεν είναι ικανοποιημένα με αυτό, διότι ορισμένα κράτη-μέλη βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση. Θα συνοψίσω την ερώτηση για να μην ξεπεράσω το χρόνο μου. Η Επιτροπή είπε ότι τα κονδύλια θα δοθούν ε, σύμφωνα με ιστορικά κριτήρια στα κράτη-μέλη, αλλά πολλά κράτη-μέλη πιστεύουν ότι αυτό είναι άδικο και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο επιμένουν για την απελευθέρωση της αγοράς. Δεν νομίζετε ότι χρησιμοποιώντας ιστορικά κριτήρια διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Νεβιτσεύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. για το 2010 υπάρχουν ορισμένα ε, σημάδια βρίσκουμε όσους υποφέρουν από τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης θα ήθελα οι απαντήσει αυτέ να μην είναι αποτέλεσμα μια συγκυρία, αλλά μια μικροπρόθεσμη στρατηγική για την αποκατάσταση και σταθεροποίηση του τομέα αυτού στην Ευρώπη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα μέτρα που θα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη και θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σα πάνω στο γεγονό ότι οι αλλαγέ στον κανονισμό 12-14 μόνο εν μέρη θα εφαρμοστούν από την Βουλγαρία. Θα πρέπει να γράψουμε λοιπόν ότι οι δυνατότητε, αλλαγής των ποσοστώσεων θα γίνουν κατά τη διάκριση των κρατών μελών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την δυνατότητα να εξαγοράσουν ποσοστώσεις ανάλογα με τα εθνικά αποθέματα. Δεν μπορούμε να αποθηκεύουμε το γάλα ε, της, ε, των αγροτών ε, διότι μετά το 2013 δεν θα είναι πια ανταγωνιστές οι Βούλγαροι, ανταγωνιστικοί οι Βούλγαροι αγρότες. Ευχαριστούμε κύριε Νεντέλτσεβα. Για ένα λεπτό τώρα ο επόμενος. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, βέβαια και χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση για να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι ακόμα και η Πολωνία. Όμως να μην ξεχνάμε ότι εδώ μιλούμε για χρήματα και το θέμα είναι πώς θα δαπανηθούν αυτά τα χρήματα, πώς θα μοιραστούν, θα φτάσουν σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο, αυτοί οι οποίοι ταλανίζονται περισσότερο από την κρίση. Εγώ δεν θέλω όλοι να πάρουν από λίγο, γι' αυτό δεν βοηθά κανέναν. Επίσης, καλό είναι πριν σχεδιάσουμε το μέλλον να μελετήσουμε την ιστορία, διότι πριν από κανένα 1,5 χρόνο ήταν μια χαρά οι τιμές για το γάλα. Και τότε έπαιρναν επιδοτήσεις τόσο ώστε να εξυγχρονιστεί ο κλάδος θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον επί τη βάση των λαθών που κάναμε στο παρελθόν, διότι έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν. Άρα να κάτσουμε για να σχεδιάσουμε το πώς θα αναπτυχθεί ο, ο κλάδος. Το να δαπανούμε χρήματα για άμεσες ενισχύσεις σου πρώτη ανάπτυξη της Πέτρου ε, ε, και τέτοιου είδους ρυθμίσεις ποστός δεν λέει τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε. Και τώρα για ένα λεπτό έχει ο κύριος Σιγιάσκη το λόγο. Κύριε Επίτροπε, μία ερώτηση. Τα 280 εκατομμύρια ευρώ προς τι θα χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω αναδιάρθρωση. Περίπου 20 κρατημέλη επιθυμούν μία ένεση στην αγορά τους. Εγώ θα ήθελα τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για μηχανισμούς στήριξης. Δεν νομίζω <clears throat> ότι οι γεωργοί μπορούν να συνεχίσουν τον εξυγχρονισμό. Δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν δάνεια. Δεν είναι κατάλληλη χρονική στιγμή για επενδύσεις. Τα 280 εκατομμύρια ευρώ σημαίνουν 2 ευρώ ανατόνο παραγόμενου γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν επιθυμεί να μειώσει την παραγωγή μέσα από το σύστημα της διαχείρισης ε, των ποσοστώσεων. Αλλά τελικά ίσως ε, συμβεί αυτό που συνέβη με τη ζάχαρη. Να καταλήξουμε δηλαδή με έλλειψη γάλακτος. Πιστεύετε εσείς ότι είναι κατάλληλη χρονική στιγμή για να μειωθεί η παραγωγή γάλακτος και σιτηρών. Εγώ δεν νομίζω. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Ντόρφμαν. Κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητή κυρία Επίτροπε, χαίρομαι πάρα πολύ κυρία Επίτροπε που εσείς λίγες μόνο εβδομάδες μετά την ε, έγκριση του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το γάλα μας καταθέτετε μέτρα για να καλύψετε τα αιτήματά μας. Όσον αφορά ε, το άρθρο 186, συμφωνώ με την πρότασή σας, συμφωνώ και με το χρονικό περιορισμό που προτείνετε που μου μοιάζει πολύ λογικός. Και εγώ τάσομαι υπέρ της διαφοροποιημένης προσέγγισης των ποσοστώσεων. Ε, αλλά ε, όσον αφορά την επαναγορά των ποσοστώσεων, αυτό με προβληματίζει. Εσείς μήνες ολόκληρους μας λέγατε ότι η τρέχουσα κρίση δεν προκλήθηκε από το σύστημα των ποσοστώσεων. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η πρόταση που κάνετε της ε, ανάκτησης των ποσοστώσεων για μένα δεν είναι λογική. Και θέλω να σας πω ότι και τελικά αυτό δεν μπορεί να είναι το τέλος της ιστορίας. Πρέπει να θεσπιστούν επιπρόσθετα τα μέτρα και για άλλε περιοχές, κυρίως για τις ορεινέ περιοχές, όπου δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική λύση παρά από το να ε, παράγουν γάλα. Τελευταίος ο η κυρία Τέστιντερ, για ένα λεπτό. Αξιότιμη Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 280 εκατομμύρια. Ελπίζω τα χρήματα αυτά ε, στην, στον, στην πλήρη έκτασή τους να δοθούν στους αυστριακούς παραγωγούς που τα χρειάζονται πάρα πολύ επιγόντως. Γνωρίζετε την κατάσταση στις ορεινές περιοχές και την κατάσταση με τις μικρές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ε, η Αυστρία είναι κατά ε, της εκπνοής των ποσοστώσεων. Εσείς είπατε την άποψή αλλά εμείς προσπαθούμε να προετοιμάσουμε τους γεωργούς μας ε, όσο καλύτερα γίνεται. Την ε, πρότασή σας για το πρόγραμμα εθελοντικής ανάκτησης στις ποσοστώσεων. Δεν το κατανοώ. Εάν το πράξουμε αυτό, τότε θα προκύψει ε, η αύξηση της τιμής των ποσοστώσεων που θέλουμε να αφήσουμε να εκπνεύσουν. Και πώς θα το εξηγήσουμε αυτό στους αυστριακούς παραγωγούς. Ευχαριστούμε. Η κυρία Επίτροπος έχει το λόγο. Η κυρία Φίσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχοντας ακούσει πολύ προσεκτικά τους ε, βουλευτές εδώ σήμερα. Ε, δημιουργείται σε κάποιον που δεν ξέρει τουλάχιστον εντύπωση ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε. Προς Θεού. Προς Θεού. Ορισμένοι τουλάχιστον από εσά γνωρίζετε τι γίνεται από τον Ιανουάριο φέτος που ξεκινήσαμε με ιδιωτική επαθυματοποίηση παρέμβαση, εξαγωγικές επιστροφές Έχουμε λάβει πολλά και διάφορα μέτρα από την αρχή του έτους. Τα νέα μέλη αυτού του Κοινοβουλίου θα πρέπει να μελετήσουν καλύτερα τα πράγματα για να γνωρίζουν τι γίνεται όχι μόνο από τότε που ανέλαβαν αλλά και από τον Ιανουάριο που έχουμε αρχίσει εμείς τη δουλειά. Τώρα, για τις συγκεκριμένες δύο προτάσεις που έγιναν το νέο το καθεστώς αυτό δεν είναι νέος δεν είναι νέο, υπάρχει και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν εξαιρετική βοήθεια δηλαδή τα κράτη μέλη είναι μια προσφορά, γι' αυτό δεν είναι υποχρεωτική υπάρχει η δυνατότητα να βοηθήσουν με την εξαγορά της ποσόστοσης που διατηρείται στο εθνικό αποθεμά και μετά επαναδιαφέρει νέμεται, επανακατανέμεται για την ακριβή. Αυτό ήταν ένα κομμάτι της συζήτησης. Το άλλο κομμάτι που ήταν και μακράν το πιο ενδιαφέρον είναι το 186. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πω ότι ο λόγος για τον οποίο βάζουμε τα γαλακτοκομικά προϊόντα στο άρθρο 186 είναι ότι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αντιδρούμε ταχαίως δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί το γάλα να μην συμπεριληφθεί στο άρθρο 186, όπως συμμετέχουν, όπως συμπεριλαμβάνονται και πολλοί άλλοι τομείς, όπως το κρέας ας πούμε, το είπα και πριν. Όσοι φοβούνται ότι με αυτή την κίνηση δίνουμε λευκή επιταγή στην Επιτροπή που μπορεί να κάνει πια ό,τι θέλει, λέγουν ορισμένοι, να σημειώσω ότι το 186, το άρθρο 186 εκφύσεως εξορισμού είναι ένα σύστημα που προβλέπει ελέγχους, που προβλέπει συζητήσεις, που προβλέπει διαχειριστικές επιτροπές. Δεν πρόκειται λοιπόν για λευκή επιταγή. Τώρα, λέτε μικρότερη, βραχύτερη περίοδος, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια. Το άκουσα. Δεν συμφωνώ, αλλά το άκουσα και το λαμβάνω υπόψη μου. Τώρα, αναφέρθηκαν και πολλά ανακριβή πράγματα. Τα 280 εκατομμύρια δεν είναι για αναδιάρθρωση, το είπε κάποιος. Είναι η δυνατότητα που έχουμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα όταν οι διατυπώσεις ολοκληρωθούν και όταν γίνει δεκτό αυτό από τη συνάντηση της ομάδας ΕΚΦΙΝ τον Νοέμβριο όταν υπογραφεί και ο προπολογισμό ε, για το 2010 θα μπορέσουμε να δράσουμε άμεσα. Αλλά αν δεν βάζαμε το γάλα στο άρθρο 186 δεν θα είχαμε τη δυνατότητα ακόμα και με όλα αυτά να δράσουμε άμεσα. Από τον εθνικό αυτό φάκελο το κράτος μέλος καταβάλει το ποσό που του αναλογεί στους πλέον ευπαθείς. Τώρα, αν αρχίσουμε αενάως και ατέρμονα να συζητάμε το θέμα της παραγωγής και της κατανομής αυτής, θα ακουστούν πολλές ευφυΐσιμες σίγουροι ιδέες, αλλά κοινό παρανομαστή και λύση δεν θα μπορέσουμε να βρούμε. Γι' αυτό εμείς αποφασίσαμε ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι και τώρα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Τώρα, οι ενώσει παραγωγών οι ενώσεις παραγωγών είναι μια εξαιρετική και θα έλεγα και απαραίτητη λύση. Όταν συζητούσαμε πέρσι το καθεστώς για τα φρούτα και τα λαχανικά είχα πει ότι αν οι γεωργοί, αν, ξοδεύουν το χρόνο τους να πολεμάνε ο ένας τον άλλον, να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αντί να ανταγωνίζονται τα μεγάλα συμφέροντα και τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, ε, δεν θα κερδίσουν ποτέ τίποτα. Πρέπει να πορευθούν μαζί λοιπόν όλοι οι μικροί και ανεξάρτητοι γεωργοί. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να βελτιώσουν τι συνθήκες υπό τι οποίε εργάζονται. Περνάω σε άλλο θέμα. Συμφωνώ απόλυτα με τον ε, αξιότιμο, με το αξιότιμο μέλος που είπε ότι αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα ε, στον κόσμο με την ε, φτώχεια και την πείνα. Και γι' αυτό μου πληγώνει, μου, μουραγίζει ραγίζει η καρδιά όταν βλέπω να χύνονται τα γάλατα στους δρόμους. Δεν είναι αυτό που κάνει καλό στην εικόνα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Ο κύριος Μποβέ και ο κύριος Χάουσλινγκ είναι άξιον θαυμασμού ότι κατάφεραν που έμειναν στα χρονικά όρια που τους έχετε βάλει, Πρόεδρε. Βέβαια θα είχε λιγότερο χρόνο ήταν εδώ ο κύριος Μποβέ όταν ήταν προγραμματισμένος να είναι και γύρισε αργότερα. Ευφύης, ευφύης η κίνηση του την αναγνωρίζω. Ευχαριστώ Επίτροπε. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Πέμπτη για το θέμα αυτό. Η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα αύριο. 9 με 1 και 3 με 7. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί στο ε, έγγραφο συνεδρίας και στο ίντερνετ. Λύεται η συνεδρία.